El presidente. Dichiaro Κυρίσω την ε, επανάληψη της ε, συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού, ε, της, Σύνοδου, της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεκόπη τον, την 5η 17 Απριλίου. Αύριο θα ξεκινήσει η Διεθνής ξεκινησει η διεθνη ημερα που είναι αφιερωμένη στη, στα στις τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορίας.